Ε, ε, πριν περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της σημερινής της διάταξης, έχω να σας κάνω δύο ανακοινώσεις. Πρώτον, σύμφωνα με το άρθρο 216 εδάφιο 4 του κανονισμού μας, σας γνωστοποιώ ότι στη διόρθωση που έκανε χτες ε, το απόγευμα η Ολομέλεια στις 5 δεν ζητήθηκε ψηφοφορία οπότε και ε, ούτως εγκρίνεται. δεύτερη ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο